Δεν χρειάζεται μόνο έλεγχο στα σύνορα. Πρέπει να μπορούμε να αποφασίζουμε ποιο μπορεί να μπαίνει και ποιο δεν μπορεί να μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ εδώ έχουμε μια πλειοψηφία που αναζητεί απλέ λύσει και νομίζει ότι θα καλύψει τα προβλήματα με λεφτά. Ενώ τα προβλήματα στην πραγματικότητα επιδεινώνονται. Και οι νέοι δεν θα είναι έτοιμοι όταν θα ξεσπάσει νέα κρίση και αυτό σίγουρα δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. Αν θέλουμε Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στους πολίτες πρέπει τη βούληση των πολιτών να αντιλαμβάνουμε υπόψη μας στα σοβαρά και χρειάζεται να γίνει κάποια στιγμή μια σωστή συζήτηση για αυτό το θέμα. Η κυρία Βίξτρο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο την Ρομπέρτα Μέτσολα για την πολύ καλή δουλειά της. Σα ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ετών. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την πολύ καλή αυτή πρόταση. Όταν πετάω στην Ευρώπη, εγώ δεν βλέπω σύνορα. Αυτό το είχε πει ο πρώτος πρόεδρος της ελεύθερης Τσεχοσλοβακίας, ο Βάκλαβ Χάβελ. Η μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής ένταξης, η κατάργηση των εσωτερικών σύνορων, βασίζεται στο να έχουμε ισχυρά εξωτερικά σύνορα. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη οχυρό. Δεν θέλουμε να διώξουμε ανθρώπους. Θέλουμε να ελέγχουμε τις ροές των ανθρώπων που μπαίνουν και βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται ένα σωστός έλεγχος ασφαλείας, υπάρχει μια διέλευση συντεταγμένη για όλους όσους έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντα ε, ε, διεθνή προστασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ουσιών, ε, παράνομων ουσιών που δεν θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση που εγκρίνουμε σήμερα δεν πάει προς ένα πλήρες ομοσπονδιακό σύστημα. Ε, για μένα αυτό είναι ο σωστός δρόμος, αλλά έχουμε γίνεται ένα πρώτο βήμα από τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι εγώ είμαι 10 χρόνια εδώ. Είναι από τι τελευταίε μου ομιλίες ε, στο Κοινοβούλιο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλους όσους με τους οποίους συνεργάστηκα όταν τελειώνει η πολιτική η φιλία μένει και είναι μια ευκαιρία για μια νέα αρχή. Ευχαριστώ. Είστε αισιόδοξοι και καμιά φορά η, πολιτική καταστρέφει φιλίε τέλο πάντων, ελπίζω να ισχύσει αυτό που λέτε στην προηγουμένη περίπτωση. Η κυρία Φορέντζα έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 1.311 θάνατοι μόνο και μόνο το 2018. Αυτός είναι ο απολογισμός των θανάτων στη Μεσόγειο. Και εμεί συνεχίζουμε και συζητάμε εδώ πέρα για σύνορα και για ενίσχυση της πολιτικής επιστροφών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει σε ένα διαφορετικό δρόμο. Καταρχάς, θα πρέπει να κηρύξει ως μη ασφαλής τους λιμένες της Λιβύης. Το έχει κάνει αυτό επίσημη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμω υπάρχουν κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρούν ότι είναι ασφαλεί οι επιστροφέ στη Λιβύη και στι χώρε αυτέ συγκαταλέγεται και η Ιταλία αν πραγματικά θέλουμε να μας θυμόμαστε, να μας θυμάται ο κόσμος ως αυτοί που αύξαν τους θανάτους στην Μεσόγειο, τότε δεν έχουμε παρά να συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό. Το αντίθετο όμως θα έπρεπε να ελπίζουμε. Σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παραπέμπουμε στις λιβικές αρχές την όλη αρμοδιότητα και ευθύνη της έρευνας και της διάσωσης. Καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία με την αστευτική μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λιβύης. Ε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ακολουθούμε την πολιτική του Σαλβίνη. Πρέπει να είμαστε μια πολιτισμένη ήπειρο. Η κυρία Βαλέρο έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουμε την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που φεύγουν από τις χώρες τους εξαιτία ένοπλων συγκρούσεων και από ό,τι φαίνεται η τάση αυτή θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Θα έχουμε όλο και μεγαλύτερα μεταστευτικά κύματα εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε εκατομμύρια κλιματικών λεγόμενων προσφύγων. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τους 600.000 ε, πολίτες οι οποίοι θα πληγούν λόγω της αύξησης της στάθμης της θάλασσας σε διάφορες χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί θα προσπαθήσουν να έρθουν προς την Ευρώπη, όχι όλοι βέβαια, αλλά εμείς πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να έρθουν προς, την Ευρώπη. Επενδύουμε αυτή τη στιγμή τεράστια ποσά προκειμένου να τους απομακρύνουμε, προκειμένου να κρατήσουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι τα χρήματα αυτά δεν θα έπρεπε να τα δίνουμε για την απομάκρυνση των ανθρώπων αυτών, αλλά περισσότερο για τη μείωση τη φτώχεια και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσή του. Ο κύριο Κορά, όχι το λόγο τώρα για μισή λεπτό. Α το πούμε ξεκάθαρα, αγαπητοί συνάδελφοι, απέτυχε η μεταρρύθμιση του κοινού συστήματο ασύλου. Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια τίποτα δεν έγινε προκειμένου να τροποποιηθεί η Συμφωνία του Δουβλίνου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι βυθίζεται σε ένα νέο εμφύλιο πόλεμο η Λιβύη και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τι επερχόμενε μεταναστευτικέ και προσφυγικέ ζωέ από τη Λιβύη. Νομίζω ότι η Frontex αυτή τη στιγμή είναι το μόνο εργαλείο το οποίο έχει απομείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση εξωτερικεύει το, το πρόβλημα αυτό, δίνει χρήματα σε τρίτε χώρε για να κάνουν αυτέ τη βρώμικη δουλειά. Και από την άλλη η μεταρρύθμιση του Frontex συνάδει ουσιαστικά με την πολιτική αυτή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, ελπίζουμε μέσω της μεταρρύθμισης αυτής, ε, ελπίζουν ορισμένοι τουλάχιστον, να κερδίσουν περισσότερες ψήφους στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Ανταυτού όμως ε, θα έπρεπε να είχαμε περισσότερη ευρωπαϊκή ελληνική, την οποία όμως δεν θέλουν καν να ακούσουν, ούτε καν ως ιδέα, ως έννοια, ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο οι χώρε εκείνε που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και οι οποίε καλούνται να διαχειριστούν τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω επίσης ότι ε, στις ε, χώρες αυτές θα έπρεπε να τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν ακόμα και εσωτερικούς ελέγχους, τη στιγμή που τους ελέγχους αυτούς δεν μπορεί να κάνει ο οργανισμός, ο Frontex. Κανονικά η αρχή τη αλληλεγγύη υποτίθεται ότι προβλέπεται από τι συνθήκε, αλλά στην πράξη δεν ισχύει, δεν λαμβάνει χώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριος Παρά το γεγονό ότι έχει αποδειχθεί στην πράξη πω το Frontex είναι το πλέον ανεπιτυχέ πείραμα για να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να τον αναβαθμίσει και να τον μετατρέψει σε οργανισμό Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή. Ε, το αυξάνει την επιχειρησιακή δύναμη σε δέκα χιλιάδε άτομα και σε περιόδους αγρίας λιτότητα φορολογεί τους ευρωπαίους πολίτες και σπαταλά τα χρήματά τους για να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό άρα και άχρηστο οργανισμό. η αιμονή όμως και η σκοπιμότητα να αφαιρεθούν από τα εθνικά κράτη αρμοδιότητες ζωτικές για την επιβίωσή τους όπω είναι η ασφάλεια των συνόρων οδηγεί την ευρωπαϊκή ένωση να λάβει αποφάσει που αντίκειται στην κοινή λογική διότι ποιο λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο θα διαφωνήσει με την άποψη ότι η καλύτερη προστασία των συνόρων ενό κράτου επιτυγχάνεται εάν η αποστολή αυτή δοθεί στι ένοπλε δυνάμει και τα σώματα ασφαλεία του κράτου αυτού. η ορθότητα αυτή τη απόψεω έχει αποδειχθεί στην πράξη διότι όλα τα κράτη τα περισσότερα κράτη τη ευρωπαϊκή ενώσεω κλείνουν τα σύνορά του για να αντιμετωπίσουν τα ανεξέλεγκτα κύματα των λαθρομεταναστών και έτσι μεταφέρουν το πρόβλημα στα κράτη εισόδου όπω είναι η ελλάδα η οποία εάν δεν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει μόνη της να προστατεύσει τα σύνορά της ουδής μαθητευόμενος μάγος της ευρώπης θα τη βοηθήσει υπό οποιαδήποτε μορφή και όνομα και αν εμφανιστεί αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Διάς Δεμέρα τώρα έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, θέλω να συγχαρώ τη Ρομπέρτα για την καλή δουλειά της. Υπενθυμίζω όμως ότι οι πιο σημαντικέ προτάσεις του πακέτου ασύλου και μετανάστευσης ε, μένουν αυτή τη στιγμή κολλημένες στον τρίλογο. Ε, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερες δυνατότητε ε, σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή στην Οριοφυλακή και θα ψηφίσουμε υπέρ. Είναι σημαντικό να ψηφίσουμε υπέρ αυτού του εργαλείου για να υπάρχουν απαραίτητε δυνατότητε που θα εγγυηθούν μια ολοκληρωμένη διαχείριση τη μετανάστευση με αποτελεσματικότητα και με ένα υψηλό επίπεδο ασφάλεια στο ιστορικό τη Ένωση, Ταυτόχρονα θα πρέπει βεβαίω να διαφυλάξουμε την έτσι κυκλοφορία των προσώπων. Η δημιουργία ενό σώματο 10.000 ανθρώπων, η υποστήριξη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι επιστροφές ή η εντετικοποίηση τη συνεργασία με τρίτες χώρε είναι πολύ σημαντικά επιχειρησιακά στοιχεία για να εγγυηθούν μια συνεχή υποστήριξη και για τις χώρες προορισμού και για τις χώρες προέλευσης και για τις χώρες transit. Από κοινού τη Europol αυτή η νέα υπηρεσία θα είναι η λιδία λίθος που θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας στην Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε το έργο μας για να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερε επιχειρησιακέ, να δώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερε επιχειρησιακέ και δημοσιονομικέ δυνατότητε σε αυτή την υπηρεσία. Υπάρχει βεβαίω και μια δικλίδα ασφαλεία, διότι αυτή, αυτό το σώμα υπόκειται στο δίκαιο τη θάλασσα, στο διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο και στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φαγιών έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Σίγουρα χρειάζεται καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό για την καλύτερη λειτουργία του χώρου Σέγγεν, για την ε, ρύθμιση της μετανάστευσης. Χρειάζονται συμφωνίες ε, για την ε, επέκταση και ενίσχυση του Frontex. Θα ψηφίσω υπέρ. Είναι σημαντικό να έχουμε την αύξηση αυτή ε, στις 10.000 μέχρι το 2027. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν την βασική ευθύνη για τη διαχείριση των συνόρων τους και θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατέψουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων που θα επιστραφούν από τη Frontex στις τρίτες χώρες. Η συνεργασία με τρίτες χώρες ε, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νέων συμφωνιών που θα λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, προσοχή, οι νέοι κανόνες για τα εξωτερικά σύνορα δεν θα πρέπει να ισχύουν χωρίς να προσαρμοστούν και για τον ε, ευρωπαϊκό εξωτερικό χώρο. Ευχαριστώ. Ο Τσαμπάσκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σαφώς θα πρέπει όλα αυτά τα χρήματα να δοθούν στο νέο αυτό οργανισμό. Τα εξωτερικά σύνορα είναι θεμελιώδους σημασίας, προκειμένου πραγματικά να έχουμε ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χαιρετίζω την διευρυμένη αυτή αρμοδιότητα που δίνεται στο νέο αυτό Frontex, και είμαι σαφώ υπέρ τη θέσπιση του μόνιμου αυτού σώματο με επιχειρησιακή δύναμη 10.000 ατόμων. Το έχω πει πολλάκι στο παρελθόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού για να σταματήσουμε την έλευση των παράτυπων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικοί μετανάστε, οι οποίοι δεν δέχονται τι αξίε μα και τον τρόπο ζωή μα, δεν έχουν καμία θέση στι χώρε μα ούτε βέβαια και οι τρομοκράτες, ε, οι οποίοι χρησιμοποιούν πολλέ φορέ τις οδού μετανάστευση. Σα ευχαριστούμε. Ουρτασούν παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η θητεία θα περάσει στην ιστορία για την ντροπή των 18.000 νεκρών στη Μεσόγειο σύμφωνα με τη Διεθνή ε, Οργανισμό Μεταναστών και το τελειώνουμε τη θητεία με το χειρότερο τρόπο με, τον, με την μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, του κανονισμού του ασύλου που έχουν μπλοκαριστεί και έχουμε τώρα αυτόν τον νέο κανονισμό για μια ακτοφυλακή στην με δισεκατομμύρια που διατίθενται χωρίς να υπάρχει ένας μηχανισμός που να διαφυλάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς μια σαφή εντολή για την διάσωση στη Μεσόγειο όπως έχει ζητήσει αυτό το κοινοβούλιο στη διαπραγμάτευσή της και στην πραγματική εντολή της το έχουμε ζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν οι κυβερνήσει τελικά ποινικοποιούν τις ΜΚΟ όπως το Open Arms που δεν μπόρεσε, μπόρεσε να ε, φτάσει να, να, να πιάσει λιμάνι στη Βαρκελόνη ε, ποινικοποιούμε λοιπόν τις ΜΚΟ ε, και δεν γίνεται αναφορά σε μια δημόσια προσπάθεια διάσωσης. Είναι πραγματικά μια ντροπή. Στη νέα θητεία θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκάλ έχει, δύο, έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η Frontex τη θεωρία ε, θα μπορούσε να προστατεύσει τα σύνορα της Ένωσης όμως είναι ευθύνη των κρατών μελών κυρίως αυτό. Η ενίσχυση λοιπόν της, ε, των αρμοδιοτήτων της Frontex ε, είναι κάτι που θα μπορούσε να διακυβεύσει την ε, κυριαρχία των κρατών μελών. Δεν πρέπει να παρεμποδιστούν τα κράτη-μέλη από το να προστατεύσουν τα σύνορά τους. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν συνεργασία. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό στην πράξη. Ανησυχούμε, διότι η συμφωνία που επετεύχθη δεν επιτρέπει στην Frontex να έχει την υποστήριξη των αρχών ε, σε τρίτες χώρες όπως τη Μακεδονία και δεν θα μπορεί να βοηθήσει για την επιστροφή των πάνω μεταναστών. Εμείς θέλαμε πάντα να υπάρξει μια ενίσχυση ε, των συνόρων και έχουμε καταφέρει εμεί να προστατεύσουμε τα σύνορά μα χωρί την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Η Ουγγαρία όμω δεν είδε ποτέ λεφτά για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κυρία Γκυλιόμ. Ίσως να ήταν τελικά απαραίτητο να ενισχυθεί η υπηρεσία Frontex, διότι τα κοινά μα σύνορα πρέπει να τύχουν διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζω λοιπόν αυτή τη μεταρρύθμιση ε, τη Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή που πρέπει να συνοδεύεται όμω από το σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων όσων ελέγχονται στα σύνορα, τα εξωτερικά τη Ένωση. Θα ήθελα όμω να αναφερθώ και σε δύο παράπονα που έχω στο τέλο τη θητεία αυτή. Ε, λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε μία ε, αποστολή διάσωση. Στη γη πάνω από 1.800 ε, άνθρωποι πέθαναν το 2018. Άνθρωποι κινδυνεύει ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί με τέτοια υπηρεσία να το κάνει αυτό. Ε, εδώ και 6 μήνες οι ΜΚΟ το κάνουν αυτό ε, στην θάλασσα. Ε, κλείνουν τα σύνορα, τα κράτη-μέλη. παρόλα αυτά συνεχίζουν οι την να να περάσουν και βεβαίως υπάρχει δεύτερη μεταρρύθμιση της Frontex, ε, χωρί να υπάρχει καμιά μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά το καθεστώ ασύλου. Και γι' αυτό λυπάμαι και φταίνουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό που μπλοκάρουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, ενώ το Κοινοβούλιο έχει θέσει τη θέση του επιτάπητο εδώ και δύο χρόνια. Ευχαριστώ κυρία Τόμας, για και ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Frontex πρέπει να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Αλλά είναι λάθος η κατεύθυνση που του δίνουμε το οργανισμό αντί να εξειδικεύεται σε επίγουσες καταστάσεις ε, και γρήγορη αντίδραση, δημιουργούμε γραφειοκρατικές υπηρεσίες τώρα. Είναι αμφισβητούμενο το πόσο θα αποδώσουν. Πρέπει να λύσουμε άμεσα τα προβλήματα. Η Frontex δεν μπορεί να ε, συμμετέχει σε επιχειρήσεις από τρίτες σε τρίτες χώρες. Δεν θα μπορεί να επιστρέψει ε, από τις, βόρειες Ευρω... Ε, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, τις χώρες από όπου προέρχονται. Εμείς είμαστε καταδικασμένοι να αντιμετωπίζουμε το οργανωμένο ε, έγκλημα και την παράτυπη μετανάστευση ε, στο κατόφλι των χωρών μας, ε, ενώ θα έπρεπε να γίνεται αυτό όσο γίνεται πιο μακριά. Σας ευχαριστούμε κύριο Ραγχέλ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Πουσιάζει όμως. Η κυρία Κιέγγε για ένα λεπτό τότε παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προώθησε τη μεταρρύθμιση του κανονισμού που θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τι ιστορικέ διχόνοιε, διαπραγματευτήκαμε και καταλήξαμε τελικά σε ένα κείμενο το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να ήταν πιο φιλόδοξο, αλλά σίγουρα θα συμβάλλει το να παγιώσουμε έναν από τους τέσσερις πυλώνες που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση και αναφέρομαι βέβαια στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια στο πλαίσιο του πυλώνα αυτού καλεί την Ευρώπη να ενισχύσει τη δραστηριότητα έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Θα πρέπει προφανώ να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων. Αυτό αληθεύει. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επομένω, η υποστήριξη τη μεταρρύθμισης αυτή θα επιτύχει μόνο αν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά και αν εξασφαλίσουμε επίση τη δραστηριότητα έρευνα και διάσωση που θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και να κάνω μια έκκληση στο τέλο τη θητεία αυτή. Σα παρακαλώ πολύ, εκινήστε εκ νέου την επιχείρηση Σοφία και δώστε τι μεγαλύτερε δυνατότητε έρευνα και διάσωση. Ο κύριος Ράντεφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν πριν από πέντε χρόνια ξεκίνησα την εντολή μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την εποχή εκείνη η όλη ιδέα θέσπιση ε, αυτού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνορεφυλακής και Εκτοφυλακή ήταν ένα πολύ ασαφέ και θεωρητικό σχέδιο. Θεωρούσαμε ότι θα έβλεπε το φω τη ημέρα το νωρίτερο το 2030. Είμαστε όμω πάρα πολύ αφελεί τότε, γιατί μέσα σε ένα χρόνο είδαμε πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγε να καταφθάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασχίζοντα τα εξωτερικά μα ε, σύνορα και οι τότε συνοριοφύλακες δεν ήταν σε θέση να διχειριστούν ένα τόσο ακραίο φαινόμενο. Έπρεπε λοιπόν επιγόντως να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και συνειδητοποίησαμε ότι ο χώρο Σέγγεν είναι πάρα πολύ σημαντικός και ότι εξαρτάται πάρα πολύ από τη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων. Συνειδητοποίησαμε τότε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια των εξωτερικών της σύνορων καταρχάς και τέσσερα χρόνια αργότερα να που συζητάμε για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοροφυλακής και Εκτοφυλακής. Λέμε ότι θα εμπεριέχει και ένα μόνιμο σώμα με δύναμη 10.000 ατόμων. Συζητάμε επίση για τι νέε αρμοδιότητε του οργανισμού αυτού. Μα νομίζω ότι ο οργανισμό αυτό από μόνο του αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύη μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών, αν θέλετε, κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέκα άνθρωποι είναι στο κατάλογο για το Eye. Θα ήθελα πραγματικά να δώσω σε όλους το λόγο, όμως σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό που θα σας δώσουμε, διότι στις πέντε ψηφίζουμε και έχει υπάρχει άλλο ένα θέμα στη μέση διάταξη πριν. Οπότε σας ζητώ πολύ ευγενικά να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό της παρεμβάσης Η κυρία Σρόιντοβα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πρόταση σχετίζεται με το με πολύ μεγάλο λάθος που έγινε το 2015-2016 όταν τα εξωτερικά σύνορα της Σέγγεν δεν προστατεύθηκαν καταλήλως και υπήρξε διέλευση έως και 2 εκατομμυρίων ανθρώπων μεταναστών και προσφύγων. Κάποιοι από αυτούς ήταν όντως πρόσφυγες οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις φρικαλαιότητες του. Όμως πολλοί από αυτούς δεν ήταν επιλέξιμοι για άσυλο και θα πρέπει να επιστραφούν. Αυτό λοιπόν είναι που θα πρέπει να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εξωτερικά τη σύνορα για λόγους ασφαλείας. Όταν έχουμε εκατομμύρια ε, οι μετανάστες οι οποίοι περνούν τα σύνορα, τότε η αίσθηση της ασφάλειας χάνεται. Γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, μετά από τρία χρόνια ε, καλής λειτουργίας, η νέα αυτή υπηρεσία, λέει κυρία Πίκουλα, ε, ο κύριος Πίκουλα θα εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία εντό της Σέγγεν Καλωσορίζω λοιπόν την θέσπιση αυτής ε, της ε, ε, δύναμης. Είναι μια αντίδραση στους κινδύνους που υπάρχουν στα εξωτερικά μας σύνορα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να εξετάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία για την ε, χορήγηση ασύλου. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για το χώρο Σέγγεν, έχει να κάνει και με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Είναι καλό ότι θα έχουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Στίβενς, η κυρία Στίβενς. Κυρία, κυρία Πρό... Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, Πάντα είμαστε υπέρ του Frontex. Πρώτη φορά το 2016 ο Frontex ανέλαβε το καθήκον να παρεμβαίνει περισσότερο στις επιστροφές ε, μετά από απόρριψη ασύλου. Και τώρα ξανά υποστηρίζουμε τον Frontex. Γιατί πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Frontex έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής. Μπορεί να είμαστε αποτελεσματικοί μόνο με ισχυρά εξωτερικά σύνορα και εδώ θα μας βοηθήσει ο Frontex. Περισσότερο, περισσότεροι πόροι, προσωπικό, θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα έτσι τις προκλήσεις. Ο Frontex θα πρέπει να δραστηριοποιείται και σε μη ε, κράτη-μέλη, ε, χώρες που βρίσκονται μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Frontex θα βοηθάει στις επιστροφές από το Μαρόκο προς μια άλλη χώρα μη μέλος, την Ιγυρία για παράδειγμα, τον Ήγηρα. Αυτό δεν μπορούσαμε, δεν το κάνουμε. Είχαμε χάσει αυτή τη δυνατότητα στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Να ε, πω ότι λυπάμαι ότι σε σημαντικό θέμα που ε, χιλιάδες ζωές εμπλέκονται και εκατομμύρια ε, ευρώ ε, δεν ε, γίνονται τακτές οι ερωτήσεις και δεν γίνεται καλή συζήτηση. Η λύση είναι το κράτος δικαίου. Αν, ο κόσμος, ε, ε, αν κάποιος επιδιώξει να μπει στην Ένωση παράνομα, θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός κανόνας που θα λέει «Παρακαλώ, λυπάμαι, πρέπει να πάτε πίσω». Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει και νόμιμη οδός για την ε, αίτηση ασύλου γιατί όλα τα πολιτισμένα κράτη δέχονται το δικαίωμα του ασύλου για αυτούς που διώκονται. Το κράτος δικαίου είναι το βασικό. Τα 11 δις ευρώ και οι έξτρα πόροι και η γραφειοκρατία θα βοηθήσουν ε, ε, να λύσουμε το πρόβλημά μας, ε, ενώ ένας πρακτικός κανόνας θα ήταν καλύτερος. Μπόκοβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση Βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε σε μια συμφωνία όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, προκειμένου να έχουμε ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα στην Ευρώπη και προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο χώρος Σέγγεν. Δυστυχώ όμω δεν αντιμετωπίσαμε έτσι τα πράγματα του 2015. Επιτέλου όμω, τρία χρόνια μετά, συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την παράτυπη μετανάστευση και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποια βήματα ακόμα. Η εντολή του Frontex θα πρέπει να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, να μπορεί να περιλαμβάνει και τις επιστροφές από τρίτη χώρα προς τρίτη χώρα. Στη Σλοβενία το 2015 είχαμε σε καθημερινή βάση χιλιάδες διελεύσεις των συνόρων μας και είδαμε ότι η τάση είναι ανωδική και τους τελευταίους μήνες και δεν νομίζω ότι πρόκειται να τροποποιηθεί πολύ στο μέλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι έρχονται από τη Βοσνία ή τη Σερβία θα, μπορούν να, θα πρέπει να μπορούν να επιστρέφονται χάρη στο Frontex. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι Ευρω... Ευρωπαίος Σοσιαλιστής Ισπανός. Είναι πολύ καλή η στόχη ενό στόχου ελεύθερης, ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ε, ε, έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, και σε αυτό θα μας βοηθήσει η ακτοφυλακή, η συνοριοφυλακή ευρωπαϊκή με μια ε, νέα δυνατότητα 15.000 ε, ε, ανθρώπους με σημαντική χρηματοδότηση. Εμείς οι σοσιαλιστές ε, συνεισφέραμε στη βελτίωση του κειμένου με τροπολογίες για να μην υπάρξουν επιστροφές σε τρίτες χώρες και να το συνδέσουμε με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το χάρτη των θεμελιώδων δικαιωμάτων που ισχύει. Όμως, πρέπει να ξέρετε ότι είναι αρκετά πικρό, πικρή η τελική γεύση, διότι υπάρχει τελικά μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και λιγότερη στον ανθρωπισμό. Στα νότια σύνορα της Ένωσης βρίσκεται η Ισπανία ε, και το πακέτο για το άσυλο ε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Το κανονισμό του Δουβλίνου επίσης είναι μπλοκαρισμένος στο Συμβούλιο. Αυτά μένουν να γίνουν από το επόμενο κοινοβούλιο. Ο κ. Μαριάς έχει το λόγο, παρακαλώ. για άλλη μια φορά θέλω να μεταφέρω την κραυγή αγωνίας των κατοίκων των νησιών του αιγαίου για τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές και κυρίως το μεγάλο αριθμό παρανόμων μεταναστών οι οποίοι εισραίουν στην ελλάδα. πρόσφατα έγινε και εκδήλωση διαμαρτυρίας στην σάμο γιατί πλέον οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. πιστεύω ότι ο ρόλος της frontex πρέπει να βελτιωθεί να μπορέσει πραγματικά να κάνει σοβαρή δουλειά στα θέματα που αφορούν την φύλαξη των συνόρων όχι μόνο στα θαλάσσια σύνορα γιατί βλέπουμε πλέον μεγάλη έλευση και από τη μεριά των χερσαίων συνόρων την περιοχή του εύρου. επομένως εδώ πρέπει να υπάρξει πολύ συγκεκριμένη βελτίωση της δουλειάς που κάνει η ίδια η frontex αλλά και στην περιοχή της Υπήρου, που υποτίθεται υπάρχει η frontex στα σύνορα ελλάδος αλβανίας και από εκεί έχουμε εισρωή κακοποιών οι οποίοι πραγματικά ληστεύουν τα παραμεθόρια χωριά. ευχαριστώ. Ποσπισίλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Παίρνω και εγώ το λόγο στα πλαίσια αυτής της συζήτησης για να χαιρετήσω την πρόταση την οποία συζητάμε και είμαι πεπισμένος ότι η έγκριση της πρότασης αυτής, η έγκριση του προτινόμενου αυτού κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοροφυλακής και Εκτοφυλακής θα αποτελέσει πολύ θετικό βήμα. Χρειάζεται σαφώς μία ενδιάμεση περίοδος προσαρμογής, αλλά πιστεύω ότι αν έχουμε ξεκάθαρους κανόνες για, τους, για τα εξωτερικά σύνορα, θα πρέπει να έχουμε παραπάνω ακόμα εργαλεία και μέσα, προκειμένου να καταφέρουμε να αποτρέψουμε και να προλάβουμε μελλοντικέ μεταναστευτικές και προσφυγικές κρίσεις. Πέρα δηλαδή από τα εργαλεία για την προστασία με των εξωτερικών σύνορων, θα πρέπει να προβλεφθούν και άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα το Ταμείο που έχουμε αυτή τη στιγμή για την Αφρική, όπου βοηθάει, θα πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον στο να επιληθούν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Τα προηγούμενα πέντε χρόνια έμαθα για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό από πρώτο χέρι. Πήγα στο Καλέ, πήγα στο Παρίσι, εργάστηκα για μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Με κάθε ευκαιρία άκουγα ανθρώπους που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν λόγω μιας μη βιώσιμης ζωής της πατρίδα τους. Έχουμε τραγική κατάσταση. Ο κόσμος ρισκάρει να πνιγεί στις θάλασσές μας για να αρχίσει μια καινούρια ζωή εδώ στην Ευρώπη. Πολλά στοιχεία χαιρετίζω. Ε, χαίρομαι που ο οργανισμός θα προλαμβάνει τους πνιγμούς. Όσοι διασώζονται θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Ε, και με τις τρίτες χώρες πρέπει να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πέρα από αυτά πρέπει να αναλάβουμε ευθύνη και να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα και τις θερήσεις που είναι τόσο πολλές ώστε να κάνουν τον κόσμο να αναλάβουν ένα επικίνδυνο ταξίδι και να φύγουν. Πρέπει να ε, προστατεύσουμε τους ευάλωτους, να προασπίσουμε τις αρχές μας και να παρασταθούμε σε ανθρώπους που θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς αν ήταν αλλιώς οι συνθήκες. Συνάδελφοι, ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση. Αναμφίβολα, μία ισχυρή και ε, συνεκτική ένωση μπορεί να λειτουργήσει με έλεγχο συνόρων. Το Είναι σημαντικό το θέμα. Δείτε την Κροατία. Η χώρα αυτή είχε τα πιο μακρά εξωτερικά σύνορα και έγινε προσπάθεια για τη διατήρηση και εσωτερικής ασφάλειας. Τώρα με το μόνιμο προσωπικό και την ταχεία ε, αντίδραση που υπάρχει θα ε, υπάρχει υποστήριξη σημαντική στα κράτη-μέλη σε κρίσιμες περιοχές. Επίσης, οι τρίτες χώρες, οι εταίροι, θα πρέπει να συνεργάζονται και να παρέχουν τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη για αποτελεσματική ε, εφαρμογή της ε, μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτρο, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική αυτή συζήτηση και για την υποστήριξή σας. Ε, κυρίως, ο νέος κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εκτοφυλακή Συνοριοφυλακή, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, αλλάζει τα πράγματα σε επίπεδο αποτελεσματικότητα στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά προστατεύει τα κοινά της εξωτερικά σύνορα και διαχειρίζεται τις μεταναστευτικές ροές για, τα, για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτή ήταν η φιλοδοξία μας. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο έτοιμη για το μέλλον, διότι δεν ξέρουμε τι μας ε, επιφυλάσσει το μέλλον. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και όλοι μας εδώ μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που πετύχαμε αυτό αποτελεί μέρος της κοινή μας ε, κληρονομιάς. Και η υπηρεσία αλλά και τα κράτη-μέλη θα έχουν τα εργαλεία για να προλάβουν και να απαντήσουν απέναντι στις μελλοντικέ κρίσεις τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ελπίζω ακράδαντα ότι θα υποστηρίξετε το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων κατά την ψηφοφορία αργότερα. Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρώπη νοιάζεται ότι εργάζεται προς συμφέρον τους, ότι μπορούν να εμπιστευτούν την Ευρώπη. Δεν σας αποχαιρετώ ακόμα, διότι έχουμε άλλη μια συζήτηση σε λίγα λεπτά, η οποία θα είναι και η τελευταία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Η κυρία Μέτσολα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω βέβαια και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στα πλαίσια της συζήτησης αυτής. Όντω και εγώ πιστεύω ότι αυτό ο κανονισμό θα αλλάξει ε, πολύ επικοδομητικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει τα εσωτερικά μας σύνορα να παραμείνουν ανοιχτά έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα και να ταξιδεύουν ελεύθερα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει μόνο αν προστατεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό θα καταφέρουμε λοιπόν να πετύχουμε με τον νέο αυτό κανονισμό όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοροφυλακή και Εκτοφυλακή. Με τον νέο αυτό κανονισμό βρίσκουμε επιτέλους μία λύση για πάρα πολλά εκρεμή ζητήματα. Δίνουμε τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους στον νέο αυτό οργανισμό και επίσης διασφαλίζουμε ότι ο οργανισμός αυτός θα τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα σε κάθε επιχειρησιακή του δραστηριότητα. Δίνουμε την απαραίτητη συνδρομή επίσης προκειμένου να ενισχυθεί και η συνεργασία μα με τις τρίτες χώρες. Και επίσης συμφωνούμε με μια συγκεκριμένη διακήρυξη, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί, να δύναται, να αλλάζει τον κανονισμό για την ε, διοικητική διαχείριση αυτού του οργανισμού και να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δική της πράξη να προβλέπει και την αύξηση της χρηματοδότησης για ακόμα και του προσωπικού του οργανισμού αυτού. Είχαμε δεσμευτεί ότι μέχρι το τέλο τη θητεία θα είχαμε ολοκληρώσει την σχετική νομοθετική διαδικασία. Το πετύχαμε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτή τη έκθεση. Να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό τη καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και όλου του συναδέλφου που πήραν το λόγο κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι καταφέραμε να πετύχουμε τον αρχικό μα στόχο. Θέλαμε μια θετική αλλαγή και καταφέραμε να την επιφέρουμε. Κερδίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση το σύνολό τη. Ευχαριστώ. Επαντιμίζω ότι ψηφίζουμε σήμερα από αυτού του κειμένου και τώρα θα περάσουμε απευθεία στο επόμενο σημείο τη ημέρα διάταξη. έκθεση του κυρίου Φερνάντο Λόπεθ Αλγιλάρ, κώδικα θεωρήσεων. Ο κύριο Λόπεθ Αλγιλάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κύριε Αβραμόπουλε. Ε, Γνωρίζετε ότι ήταν ε, τιμή μου που ε, εδώ και πολλά χρόνια εργάστηκα ε, πάνω στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις θεωρήσεις, τον νέο κώδικα, ε, Ευρωπαϊκό Κώδικα Θεωρήσεων που έρχεται εδώ σήμερα προς συζήτηση και τελική ψήφιση. Πολλά χρόνια σκληρής δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως όπως ήθιστε στο κοινοβούλιο αυτό τους κοιόδης εισηγητέ ε, οι οποίοι συνεργάστηκαν αποτελεσματικά και πιστά ε, για, για την εκπόνηση αυτής της νομοθεσίας και εσά βεβαίω, κύριε Βραμόπουλε, διότι παρακολουθήσατε στενά τα θέματα αυτά και ήσταν συχνά στην Επιτροπή μας ε, Ελευθερίας ε, Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης. Είχαμε πολλές ακροάσεις, συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Γι' αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που πετυχαίνει έναν κρίσιμο στόχο του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, για τον οποίο μιλούσαμε σήμερα νωρίτερα, ε, μια διαχείριση ολοκληρωμένη ε, των εξωτερικών συνόρων που εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εντό των συνόρων και που μας δίνει και τα απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία για να εναρμονίσουμε τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νόμιμους σκοπούς. Μιλάμε για τους καλόπιστους ε, ταξιδιώτες, bona fide travelers, που έρχονται για 90 έως 180 μέρες ε, στην Ευρώπη για λόγους τουρισμού, για λόγους ε, πολιτιστικούς, για λόγους αθλητικούς, για λόγους επιχειρηματικούς, για λόγους έρευνας. Όλα αυτά καλύπτονται σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Θεωρήσεων μετά από μια πολύ λεπτομερή δουλειά που έγινε, ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Έχουμε φτάσει σε μια ισορροπία λογική θα έλεγα, για να είναι ίδιες οι προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφος της Ένωσης. Με συγκεκριμένες επίσης, συγκεκριμένα τέλη για τις θεωρήσεις, σε ό,τι αφορά τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει κάποιος και βεβαίως έκανα μια μεγάλη προσπάθεια πολεμώντα θεούς και δαίμονες ε, για την διευκόλυνση, να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους καλόπιστου ταξιδιώτες. Τους ταξιδιώτες καλή την πίστη δηλαδή. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου έρχονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Έρχομαι από μια απομακρυσμένη περιοχή, τις Κανάριε Νήσου, όπου έρχονται 18 εκατομμύρια τουρίστε το χρόνο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας ε, αυτό το θέμα της διευκόλυνσης ε, της ε, εισόδου στον χώρο Σέγγεν. Μερικές τροπολογίες ήρθαν να εξορροπήσουν το κείμενο, σχετίζονται με το τέλος της θεώρησης, 90 με 180 ευρώ, με μείωση βεβαίως για τους ε, ανήλικους ε, και με εξαιρέσεις για τους ερευνητές, τους καλλιτέχνες, ε, τους αθλητές. Ε, υπάρχει ένα συμβασμός και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την υγειονομική, 15 μήνες μετά την, ίσο, την, την θέση ισχύ της νέας νομοθεσίας θα υπάρξει αναθεώρηση. Επίσης έχουμε φτάσει σε μια λογική, ένα λογικό συμβιβασμό σε ό,τι φορά τις προθεσμίες για την χωρίς τη θεώρησης, έτσι ώστε να είναι πιο απλό αλλά και πιο ε, φτηνό, διότι είναι πιο εύκολο να έρθει κάποιος να μπορεί να κλείσει το αεροπορικό του εισιτήριο νωρίτερα. Ε, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ επίσης στη σημασία της διαφύλαξης, της διευκόλυνσης, την πρόθεση της διευκόλυνσης και όχι του χαρακτήρα της ασφάλειας μόνο διότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, της παράνομης μετανάστευσης, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την νόμιμη πρόσβαση στην Ένωση. Έγινε λοιπόν μια απόπειρα να επιβληθεί μια μηχανική, αυτόματη ε, σχέση με τις επιστροφές. Εμείς όμως μιλάμε πλέον για θετικά κίνητρα προς τρίτες χώρες ε, με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την παράνομη μετανάστευση έτσι ώστε ε, να μπορέσει να εφαρμοστεί όσο γίνεται καλύτερα αυτή η νέα νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Επίτροπο, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζω τη συμφωνία επί του σημαντικού αυτού φακέλου. Για άλλη μία φορά θέλω να επενέσω τον εισηγητή, κύριο Λόπες Αγγιλάρ, και τους Κιώδης για το έργο τους στο νέο αυτό νομοθέτημα. Ο τουρισμός, τα ταξίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και όχι μόνο. Είναι περίπου το 10% του ενωσιακού ΑΕΠ. Οι επαχθείς και μακρές διαδικασίες ε, αποθαρρύνουν τους ε, επισκέπτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει λιγότερες επενδύσεις, λιγότερες δαπάνες και επηρεάζει αρνητικά η οικονομία της Ένωσης. Οι συμφωνημένες αλλαγές θα διευκολύνουν εκατομμύρια ταξιδιώτες να πάρουν θεώρηση για να ταξιδεύουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευκολύνεται έτσι ο τουρισμός, το εμπόριο και οι επιχειρήσεις η διευκόλυνση της διαδικασίας δεν σημαίνει πάσο ελεύθερο ε, ούτε πιο χαλαρή έλεγχη ασφαλείας. Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν, θα ενισχύσουν τα πρότυπα ασφαλείας, θα εντοπίζουν εκείνους που αποτελούν απειλή ή δεν δικαιούνται να εισέλθουν στην Ένωση. Ένας νέος ε, κανονισμός θα μας επιτρέπει να με τη μόχλευση της πολιτικής θεωρήσεων σε συνεργασία με μη χώρες μέλη όταν πρόκειται για την επιστροφή και επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών. Είναι Οι κανόνες περιλαμβάνουν πιο ευέλικτες διαδικασίες για επισκέπτες που εισέρχονται στο χώρο Σέγγεν. Γιατί, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, ο, η νωρίτερη ημέρα που μπορεί να κατατεθεί έτοιμα είναι τρεις μήνες πριν από το ταξίδι, ενώ οι νέοι κανόνες επεκτείνουν το διάστημα αυτό στους έξι μήνες. Η ίση μεταχείριση των ετούντων θα διασφαλίζεται επίσης. Οι συχνοί ταξιδιώτες με θετικό ιστορικό θεωρήσεων μπορεί να έχουν βίζα πολλαπλών εισόδων με σταδιακά κλιμακωτά αυξανόμενη περίοδο ε, ισχύω από ένα έτος μέχρι σιγά σιγά τα πέντε χρόνια. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και για τους ετούντες και για τα κράτη-μέλη. Παράλληλα, η εκπλήρωση των συνθήκων προϋποθέσεων εισόδου από τους ταξιδιώτες θα επαληθεύονται σε όλες τις περιπτώσεις. Σχολαστικά, μία με μια μέτρη αύξηση των τελών θεώρησης από τα 60 στα 80 ευρώ έχει επίσης προταθεί για να διασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για την ενίσχυση της ασφάλειας. Αυτή η μετριοπαθής αύξηση θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν τα σωστά επίπεδα προξενικών ε, ε, αρχών παντού. Έτσι θα βελτιωθεί η ασφάλεια και θα αναβαθμιστεί και το λογισμικό χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα για τους ετούντες θεώρηση. Για να συνοψίσω, ο νέος κώδικας θεωρήσεων της Ένωσης θα προσαρμόσει τους κανόνες τις ε, ξελισσόμενες ε, ανάγκες ε, σχετικά με την ασφάλεια θα αντιμετωπίσει την ε, παρά μετανάστευση και θα χρησιμοποιήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ελπίζω να στηρίξετε τη συμβαστική λύση που επετέθηκε και προσβλέπω στη συζήτησή μας βέβαια. Και στο τέλος των εισαγωγικών μου παρατηρήσεων θα ήθελα να ε, να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα για να πω δύο λόγια. Είναι η τελευταία σημερινή μας συνάντηση. Εμείς, όπως ξέρετε, ως Επιτροπή θα μείνουμε μέχρι το τέλος του οκτωβρίου αλλά κάποιοι από εσά δεν θα είναι μαζί μας σε λίγο καιρό από τώρα. θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες γιατί αυτά τα τεσσεράμιση χρόνια εργαστήκαμε πολύ μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης μέσα σε αυτόν τον δημοκρατικό χώρο όπου υπήρξαν θέσεις και αντιθέσεις διαφορετικές απόψεις αλλά στη τελευταία ανάλυση ο κοινός μας τόπος ήταν να δώσουμε πιστικές απαντήσεις σε μεγάλες προκλήσεις και προβλήματα όπως αυτό της μετανάστευσης και της ασφάλειας. χωρίς τη δική σας βοήθεια δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα και αν σήμερα λέμε ότι αφήνουμε πίσω μας μια κληρονομιά αυτό οφείλεται σε αυτή τη συνεργασία. θέλω λοιπόν να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να ευχηθώ σε όσους από εσάς βρεθούν στο επόμενο κοινοβούλιο να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος και με βαθιά συνείδηση του καθήκοντός τους το έργο τους αλλά και εκείνους που θα βρεθούν κάπου αλλού να θυμούνται πάντοτε ότι αυτό το πέρασμά τους από τη ζωή ήταν κάτι χρήσιμο για την πατρίδα τους και για την Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε αυτούς που βρίσκονται πίσω από την δημόσια αυτή σκηνή, τους διερμηνείς μας, που καμιά φορά τους κάνουμε και τη ζωή δύσκολη εγώ φρόντιζα τουλάχιστον να μιλάω αργά ελπίζω να το έχουν εκτιμήσει. από την άλλη μεριά όμως και τους χουισιέα, όλους αυτούς τους ωραίους ανθρώπους που καθημερινά μας συνοδεύουν στην αίθουσα και παρακολουθούν από κοντά την δουλειά μας προσφέροντάς μας τις όμορφες υπηρεσίες τους αλλά και τους φωτογράφους που αποτυπώνουν με το ταλέντο τους και την έμπνευσή τους αυτό που θα αφήσετε όλοι σε ανάμνηση του μεγάλου σας έργου στην αιωνιότητα. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω προσωπικά. Έμαθα πολλά από αυτό το περασμά μου από το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι φεύγοντας, όταν έρθει η ώρα να αποχωρήσουμε κι εμείς, θα μπορούμε να λέμε πολύ απλά ότι είμαστε κι εμείς τότε εκεί, όταν κρινόταν από τη δική μας δουλειά το μέλλον της μεγάλης μας χώρας της Ευρώπης. Κινηθήκαμε με βάση αρχές και αξίες και πρέπει να σας πω ότι αυτός εδώ ο χώρος αυτό το κοινοβούλιο μπορεί να είναι υπερήφανο με όλους τους εκπροσώπους του γιατί πράγματι αντιπροσωπεύει το βαθύτερο νόημα της ε, δημοκρατίας και των ανώτερων και ευγενών αξιών πάνω στις οποίες χτίστηκε η ευρώπη. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Νομίζω ότι ήσασταν παρόν στη δημιουργία ε, ενός ε, ολόκληρου, μιας ολόκληρης υπηρεσίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε βέβαιοι ότι και οι συνάδελφοι εκτιμούν την προσπάθειά σας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντεμόντε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω βέβαια και τον Επίτροπο για τα όσα είπε με τα οποία συμφωνώ βέβαια απόλυτα. Να ευχαριστήσω και εγώ και εσά και το προσωπικό σα, κύριε Επίτροπε. Όσον αφορά το ζήτημα που συζητάμε σήμερα, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τι εξελίξει που έχουμε, το ότι μπορούμε να έχουμε μια αναθεώρηση του κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων για να προωθήσουμε την κινητικότητα, η δυνατότητα να υποβάλει κανεί αίτηση έξι μήνε πριν το προεπόμενο ταξίδι. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι προβλέπονται χαμηλότερα τέλη θεώρηση για του νέου, το ότι μπορεί να προβλέπονται αυτή τη στιγμή πολλαπλέ θεωρήσει για του συχνού ταξιδιώτε και πιο ευνοϊκέ συνθήκε όσον αφορά του αθλητέ και τους καλλιτέχνες. Είναι κρίμα όμως ότι δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε αν μπορούμε να καταργήσουμε τον περιορισμό αυτό, τον ιδιαίτερα αναχρονιστικό, που δεν επιτρέπει σε ορισμένους καλόπισους ταξιδιώτες να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταδείξει πολλές φορές ότι υποστηρίζει τις διαμονές αυτές μεγαλύτερης διάρκειας. Το να έχουμε ένα περιορισμό 90 ημερών αυτή τη στιγμή είναι κάπως αναχρονιστικό πολιτισμοί αυτοί είχαν προβλεφθεί όταν ο χώρο Σέγγεν ήταν πολύ πιο μικρό από ό,τι σήμερα. Ο κύριο Μπέκερ τώρα έχει το λόγο. μετά από πολλέ χρονιέ καταφέραμε να εγκρίνουμε τον κώδικα θεωρήσεων. Στις διαπραγματεύσει στο ΕΛΚ μαζί με άλλου εισηγητές, συνεισηγητές, συνεργαστήκαμε και μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα, χάρη σε αυτή τη θετική συνεργασία, ήταν απόλυτα θετικό. Έχουμε μια νέα πρόταση για ένα νέο κώδικα θεωρήσεων και ευχαριστώ και το Συμβούλιο για τον θετικό και επικοδομητικό διάλογο που είχαμε. Η Ένωση στο μέλλον θα μπορέσει έτσι να ενισχύσει τις ε, σχέσεις της με τρίτες χώρες και θα επιτρέψει να αυξήσουμε και τον τουρισμό, το, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τον αθλητισμό. Έτσι επιτυγχάνουμε έναν από τους στόχους του ΕΛΚ, ε, κάτι που τελικά δέχθηκαν και οι άλλοι συνάδελφοι, την σύνδεση του κώδικα θεωρήσεων με την επιστροφή στα τρίτα κράτη. Τα τρίτα κράτη που δεν ε, συνεργάζονται δεν θα έχουν ε, δικαιώματα ε, ελεύθερης εισόδου χωρίς θεώρηση. Αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενισχύοντας την συνεργασία. Δυστυχώς αυτή η αρχή σε ό,τι αφορά και την ε, εξωτερική προστασία των συνόρων δεν υλοποιήθηκε. Και καλωσορίζω βέβαια την ενίσχυση της Frontex με προσωπικό, με χρηματοδότηση για πραγματικά αποτελεσματική συνοριοφυλακή, αλλά δυστυχώ. δεν μπορεί η Frontex να συνδράμει τι χώρε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την επιστροφή των υπηκών του. Είναι επίση λυπηρό το γεγονό ότι η Frontex ακόμα χρειάζεται την συνένεση του κράτου μέλου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την συναρπαστική αυτή περίοδο που περάσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα η κυρία Φαγιόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και χαίρομαι που βλέπω ότι μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων και με τη δεύτερη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταφέραμε να δημιουργήσουμε νέους ε, κανόνες για την θεωρήσεις. Αν εγκριθούν λοιπόν οι κανόνες αυτοί, η διαδικασία για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο απλή. Και τα κράτη-μέλη θα διατηρήσουν το βασικό τους ρόλο στη διαδικασία αυτή. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις ε, θεωρήσεις είναι το κλειδί γιατί διευκολύνει τον τουρισμό, την πρόσβαση των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργεί την εντύπωση μιας ανοιχτής, ασφαλούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω επίσης ότι αυτές οι θεωρήσεις ε, προορίζονται για τα κράτη της ε, Δυτικών Βαλκανίων. Δεν έχουν καταργηθεί τελείως, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα την καταπολέμηση του τράφικινγκ και των εγκλημάτων. Είναι τεράστιε οι ουρέ μπροστά στα προξενία για του νέου που δεν έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική για τι θεωρήσει λοιπόν αποτελεί μια πολιτική πάρα πολύ απτή, με απτά αποτελέσματα για του πολίτε. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και να είναι προ όφελο των ταξιδιωτών. Και με του νέου κανόνε που εγκρίνουμε, οι πολίτε θα είναι σε θέση να λαμβάνουν θεωρήσει με πιο γρήγορο τρόπο, να ζητούν τέτοιες θεωρήσεις ε, ε, έξι μήνες εκ των προτέρων και θα μειώνονται και τα τέλη και για τους αθλητές, τους φοιτητές, ε, τους καλλιτέχνες τα τέλη αυτά. Θα είναι χωρίς χρέωση για παιδιά. Είναι λοιπόν κλειδί αυτό. Αυτό που δεν ανέφερε ο συγητή είναι ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε αυτά που θέλαμε για τι ανθρωπιστικέ θεωρήσει. Είμαι πεπισμένη ότι αυτό θα οδηγούσε σε λιγότερη διοχέτευση, αν θέλετε, μικρότερη διοχέτευση των ανθρώπων σε μεταναστευτικές οδού. Και πρέπει να το τονίσουμε ότι χρειάζονταν αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Στίβεν, για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, συνάδελφοι, η αναθεώρηση του κώδικα για τι θεωρήσει είχε σκοπό να διευκολύνει τα πράγματα για του τουρίστε, για να ζητούν θεωρήσει. Αυτό είναι σημαντικό για την οικονομία μα και για τον τουρισμό μα. Αλλά οι θέσει μπλόκαραν επανειλημμένα την διαδικασία αυτή, γιατί θέλουν να εισαγάγουν τη δυνατότητα ανθρωπιστικών θεωρήσεων στου πρόσφυγες μέσω των προξενείων μα, όπου και αν βρίσκονται αυτά στον κόσμο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία. Η διερμηνία λειτουργεί κανονικά. Ακούτε παρακαλώ την διερμηνία, λέει η κυρία Στίβεν. Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν. Τώρα λοιπόν που επιτέλους ε, αφαιρέθηκε αυτό το εμπόδιο και μπορούμε να ψηφίσουμε την πρόταση αυτή και μπορούμε να ζητήσουμε συγκεκριμένα τέτοιες ε, συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τους τουρίστες θα μπορέσουν ακόμα πιο εύκολα να έρχονται στον, ε, στην περιοχή του Σέγγεν. Θα μειωθούν τα τέλη για την χορήγηση θεωρήσεων και τα τεκμήρια τα οποία είναι απαραίτητα μειώνονται στον αριθμό. Τα κράτη-μέλη, αν έχουν χρησιμοποιήσει ε, με σωστό τρόπο, μάλλον άτομα, οι πολίτε θα μπορούν να ζητούν και μακροπρόθεσμε θεωρήσει σε περίπτωση που έχουν ε, καλό ιστορικό. Αν οι χώρε όμω δεν ε, συνεργαστούν σε ό,τι αφορά την επιστροφή παράνομων μεταναστών, θα χάνουν τα πλεονεκτήματά τους και οι πολίτες τους θα χρειάζεται να περιμένουν μια απόφαση θεωρήσεων πιο μεγάλο χρονικό διάστημα και να πληρώνουν πιο υψηλά τέλη. Και αυτό θα οθήσει τα καθημέρινα να συνεργαστούν σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση, τη χορήγηση εγγράφων. Και επίσης δεν θα μπορούν να χορηγούνται ε, θεωρήσει μία ημέρα. Λοιπόν, ε, τέτοια λοιπόν κενά που αποδυναμώνουν το σύστημα θεωρήσεων θα πρέπει να κλείσουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η τελευταία μου παρέμβαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να σα ευχηθώ ότι καλύτερα για το μέλλον και να σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία. You're welcome. Uh, Depre. Ε, Gerard Depre, για δύο λεπτά παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, 60 εκατομμύρια. Περίπου 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, χρόνο είναι τα άτομα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό για να επισκεφθούν τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι από τι ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, και εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησεων. Άλλοι προέρχονται από 105 χώρες, κυρίω από την Αφρική, την Ασία και την ε, Λατινική Αμερική, είναι υποχρεωμένοι να έχουν θεώρηση για να μπουν στις χώρε της ζώνη Σέγγεν. Ε, η αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων που ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε ε, είναι για αυτούς ακριβώς. Θέλει να διευκολύνει τα τουριστικά και επαγγελματικά ταξίδια για τους καλόπιστους ταξιδιώτες ε, αποτρέποντας το μεγαλύτερο, στο, κατά το δυνατό, τις ε, παράτυπες ε, μετακινήσεις και μεταναστεύσεις. Η συμφωνία με το Συμφούλιο είναι καλή συμφωνία. Ε, η θεώρηση θα πρέπει να ε, ζητείται έξι μήνες πριν και να ε, εκδίδεται τουλάχιστον 15 μέρες πριν το ταξίδι. Οι πολλαπλές θεωρήσεις μπορούν να εκτείνονται για περίοδο 5 ετών και για όλα τα κράτη. Τα τέλη θεωρήσεων που δεν έχουν τροποποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια θα αυξηθούν από 60 στα 80 ευρώ για τους ενήλικους